προκειμένου να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η νέα εμπορική πολιτική στο μέλλον. Χθε είχαμε μία επικοδομητική συζήτηση για το ζήτημα αυτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη το εργαστήριο που είχαμε χθες για την έκβαση των συζητήσεών μας. Uh, uh, uh, contact with most of the issues involved in this dossier. Και καλύψαμε και πολλά επιμέρους ε, ζητήματα στα πλαίσια της συζήτησης. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον Τανιέλ Κάσπαρη... που θα μας μιλήσει για την έκθεσή του αυτή, την οποία την έχετε και μπροστά σας. Έχετε το λόγο κύριε Κάσπαρη. Ähm, σας ευχαριστώ πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε σήμερα την ευκαιρία να αναφερθώ σύντομα στην έκθεση αυτή. Πριν από μερικούς μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την μελλοντική της στρατηγική όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για την εμπορική πολιτική. Θεωρώ ότι η προσέγγιση είναι πολύ θετική, καλύπτει τα επόμενα χρόνια Ξέρουμε βέβαια ότι ε, η εμπορική πολιτική είναι μια πολιτική η οποία είναι ιδιαίτερα μακροπρόθεσμη. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλέ εμπορικέ διαπραγματεύσει οι οποίε ε, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρε. Έχουμε δει ότι για παράδειγμα ο κύκλο διαπραγματεύσεων τη Δόχα έχει ήδη διαρκέσει 10 χρόνια. Επομένω, κάθε φορά που μιλάμε για εμπορική πολιτική, για στρατηγική για την εμπορική πολιτική, θα πρέπει να ταινίζουμε το μακρινό μέλο, δηλαδή να δούμε πώ θα δημορφωθεί ο κόσμο τα επόμενα 20-30 χρόνια. Αυτό το οποίο απουσιάζει από το έγγραφο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι το τι μορφή θα έχει πάρει η οικονομία στον κόσμο τα επόμενα 15 με 20 χρόνια. Σίγουρα είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή να γνωρίσουμε ακριβώ πώ θα διαμορφωθούν τα πράγματα τα επόμενα 15-20 χρόνια, αλλά θα μπορούσαμε τουλάχιστον να δούμε ποιε είναι οι γενικότερε τάσει που αναδύονται. αν έχουμε μια αύξηση του ΑΕΠ 5-6% ετησίως στην Ινδία, την Κίνα και άλλες ε, χώρες, ξέρετε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα όσον αφορά την οικονομία και πώς θα επηρεαστεί και στο μέλλον η εμπορική πολιτική. Θεωρώ λοιπόν ότι η ευρωπαϊκή πολιτική δεν έχει αντιμετωπίσει καθόλου το ζήτημα αυτό των μελλοντικών δηλαδή εκτιμήσεων. Δεύτερον, Γίνεται συνεχώς λόγος για την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν επιτυγχάνουμε τα ευκταία επίπεδα. Θα πρέπει όμως να δούμε πώς θα εξελιχθεί η οικονομική ανάπτυξη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να γίνεται λόγος και στο έγγραφο αυτό. Ζήτησα λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί πάλι με την μακροχρόνια εξέλιξη της εμπορικής πολιτικής εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να γνωρίζουμε επίσης πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τα επόμενα 45 χρόνια, αλλά όχι μόνο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε πώς θα εξελιχθούν και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν ολοκληρωθούν, για παράδειγμα, οι κύκλοι διαπραγματεύσεων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Επίσης, Λέω στην έκθεσή μου ότι η εμπορική πολιτική δεν θα πρέπει να αποτελεί αυτό σκοπό, αλλά να συνδυάζεται με άλλους στόχους, με άλλες πολιτικές. Θα πρέπει, για παράδειγμα, στην Ευρώπη να καταβάλουμε προσπάθειες προκειμένου να ενημερώνται σωστά οι πολίτες για την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δικαιολογημένες ανησυχίε που έχουν ορισμένοι πολίτες, εκφράζουν ανησυχίε αυτές, αλλά δεν απαντώνται από τα αρμόδια όργανα ενδιαφέρονται για την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τι δυνατότητε οικονομική ευημερία, για τη δυνατότητα δημιουργία θέσεων εργασία, Πρέπει να έχουμε λοιπόν μια πολυμερή προσέγγιση και να καταφέρουμε να ενισχύσουμε την θέση μα και στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Πρέπει να γνωρίζουμε στα πλαίσια των διεθνών διαπραγματεύσεων ποιοι είναι οι συνομιλητέ μα και πώ διεξάγονται αυτέ οι διαπραγματεύσει. Πολύ συχνά στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που γίνονται για συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών δεν εκπροσωπούνται απαραίτητα τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητάμε επίση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα συζητήσει που έχουμε με του σημαντικού μα εμπορικού εταίρου. Ηνωμένε Πολιτείε, Ρωσία, Ιαπωνία. Έχουμε έναν συνεχή διάλογο με τις χώρες αυτές, χωρίς όμως να έχουμε καταλήξει σε κάποια επικοδομητικά αποτελέσματα. Δεχομένως θα πρέπει η στάση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι πιο επιθετική. Θέλουμε πιο ανοιχτές αγορές, θα πρέπει να μπορούμε να αποφεληθούμε κι εμείς περισσότερο από την οικονομική ανάπτυξη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει βέβαια να υπεραμεινθούμε και της δικής μας εμπορικής πολιτικής. θα πρέπει να μας απασχολήσει και το ζήτημα των υπηρεσιών όλο και περισσότερο. Έχουμε πολλά βιομηχανικά προϊόντα, προϊόντα υψηλή τεχνολογία, τα οποία εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση παγκοσμίω. Τα προϊόντα αυτά και οι υπηρεσίε αυτέ, μάλλον τα προϊόντα αυτά βασίζονται σε πολύ σημαντικέ υπηρεσίε, χρηματο, χρηματοοικονομικές υπηρεσίε ε, υπηρεσίες ασφάλειας, ασφάλισης και Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίσουμε πώ εξελίσσονται γενικότερα οι υπηρεσίε αυτέ παγκοσμίω. Θα πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί περισσότερο πώς ρυθμίζονται οι υπηρεσίες αυτές τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει και ένα άλλο κεφάλαιο, η καταπολέμηση της φτώχειας, καθώς επίσης και η ανάπτυξη, οι συμφωνίες οικονομικής, μάλλον οι συμφωνίες αναπτυξιακής βοήθειας, όλες οι ρυθμίσεις και συμφωνίες που υπάρχουν όσον αφορά τις προτιμησιακές συμβάσεις που έχουμε με τρίτες χώρες και να ασχοληθούμε επίσης και με τα δασμολογικά ζητήματα. Το γεγονός ότι ε, το ζήτημα της ε, καταβολής των δασμών αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα, αλλά η συγκέντρωση των δασμών αυτών, η συλλογή των δασμών αυτών γίνεται ε, αποσπασμένη μεμονωμένα από κάθε κράτος μέλος σε εθνικό επίπεδο. ακούμε όλο και περισσότερο ότι ε, υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες είναι σε θέση να επιλέγουν συγκεκριμένα αεροδρόμια εισαγωγής και εξαγωγής για τα προϊόντα. Επιλέγουν ουσιαστικά τα αεροδρόμια αυτά τα οποία επιβάλλουν χαμηλότερους δασμούς. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό, να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Προσπάθησα να συμπεριλάβω όλα αυτά τα ζητήματα στο σχέδιο έκθεσης και Προφανώς ε, περιμένουν να κάνουν προτάσεις και οι συνάδελφοι αν πιστεύουν ότι υπάρχουν κάποια σημεία πρέπει να βελτιωθούν Είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια να έχουμε κατά νου ότι μιλάμε για μια νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να επισέλθουμε σε πάρα πολλέ λεπτομέρειε. Δεν θα πρέπει να γίνονται πολλέ επιμέρου αναφορέ σε κάθε διαφορετική FTA. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πάντα κατά νου ότι μιλάμε για μια γενικότερη κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για την εμπορική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση σας δόθηκε την περασμένη Πέμπτη από τη Γραμματεία, το σχέδιο έκθεσης τουλάχιστον. Νομίζω ότι θα πρέπει να μετατοπιστεί όμως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των τροπολογιών να περάσει δηλαδή στην επόμενη, την ερχόμενη πέμπτη, την πέμπτη της επόμενη εβδομάδας. Πολλοί συνάδελφοι θα είναι στη Γενέβη και θα πρέπει να έχουν τον απαραίτητο χρόνο να μελετήσουν την έκθεση αυτή και να υποβάλουν τροπολογίες εφόσον το επιθυμούν. Σας ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω σε στενή συνεργασία τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Σας ευχαριστώ για την ε, ξεκάθαρη εισήγησή σας και την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης. Θα πρέπει ωστόσο να διαπιστώσουμε πως δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Παρότι είναι πάρα πολύ σημαντική η σημερινή συζήτηση, αυτό εδώ είναι το σημαντικότερο έγγραφο που έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμή. Με πάση περιπτώσεις, ε, ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τους ε, λίγους ε, που φρόντισαν να έρθουν. Κύριο Μάρτιν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, συμφωνώ. Είναι σημαντική έκθεση για την Επιτροπή μας και θέλω να ευχαριστήσω τον Ντάνιελ για την πολύ συνεπή και λογική απάντηση του Ντάνιελ στην ε, πρόταση της Επιτροπής. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις δυσκολίες της παγκόσμιας ευρωπαϊκής στρατηγικής, αλλά ταυτόχρονα και την παρουσίαση μιας στρατηγικής πολιτικής της Ευρώπης για την εμπορική πολιτική. Το εμπόριο, όπως σωστά είπε και ο Ντάνιελ και το τόνισε, δεν είναι αυτός σκοπός αλλά οι ορισμένε προποθέσει μπορεί να αποτελέσει κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη και άρα να οδηγήσει στη βελτίωση των συνθηκών ζωής ε, τις οποίες έχουμε συνηθίσει. Επίσης το εμπόριο μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στις ε, σε κοινωνικές προδιαγραφές, προδιαγραφές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και περιβάλλοντος και το Κοινοβούλιο έχει πρόσφατα αποφασίσει μέσω της έκθεσης ΑΕΦΗ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνική πολιτική ότι αυτά θα εντάσσονται στην εμπορική πολιτική. Επιπλέον κάτι που τόνισα στην γνωμοδότηση της Υποεπιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα βέβαια ο Ντάνελ είπε ότι δεν θέλει να επεκτείνει την έκθεση του υπερβολικά όμως αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι το σχέδιο GSP SIN. Ε, Γιατί θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το ρόλο αυτού του τύπου των συμφωνιών. Και νομίζω πως η εποπτεία του προγράμματος GSP θα πρέπει να ενισχυθεί και η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να παίξει πιο δραστηριό ρόλο, πιο ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση της εφαρμογής αυτού του προγράμματος, να φροντίζουμε τις παραβιάσεις, να, ε, να, να, περιορίζουμε μάλλον και να εφαρμόζουμε τις εμπορικέ αυτές προτιμήσεις σε σχέση με τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα, σε σχέση με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, φυσικά είμαι ευτυχής που δημιουργήθηκε η συμβουλευτική ομάδα ε, και θα ήθελα να ξέρω αν η Κομισιόν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει αυτού του είδους το μοντέλο για να φτιάξει άλλες παρόμοιες συμβουλευτικές ομάδες και να δούμε κατά πόσο η σχετική ομάδα για την Κορέα έχει προβεί σε κάποιες συστάσεις. Θα ήθελα να τα δω αυτά. Και φυσικά η σχετική συμφωνία ε, περιλαμβάνει και ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά θα ήθελα να είναι καλύτερα δεσμευτικό και όχι προαιρετικό. Να έχουμε δηλαδή συμμεταχείριση με τις εμπορικές πτυχές της ε, εμπορικής συμφωνίας και θα κάνω σχετική τροπολογία. Εν γέννη όμως ημερίζομαι τα συμπεράσματα του Ντάνιελ ότι Το καλύτερο θα ήταν ε, να ολοκληρωθούν εσίως οι διαπραγματεύσεις του γύρω της ε, ε, ανάπτυξης, αλλά πιστεύω πως θα πρέπει να συνεχίζονται και οι διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις και συμφωνώ ότι αν θέλουμε να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 ενώ το Global Europe δεν το κατάφερε, θα πρέπει να δώσουμε ένα σωστό πλαίσιο για την εμπορική πολιτική για τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. ο Σερ Καμάλ. Σας ευχαριστώ. Όπως και ο προηγούμενος ομιλητής, ε, καλωσορίζω την έκθεση του Ντάνιλ και εντυπωσιάζομαι για το πόσο σύντομη ε, την έχει κάνει, παρότι έχει να καλύψει τόσο πολλά ζητήματα που καλύπτουν και άλλες επιτροπές. Τώρα, στο μυαλό μου έχω 12 παρατηρήσεις, δεν θα σας αναφέρω όλες. Ε, μην ανησυχείτε, αλλά νομίζω πως ένα θέμα που πρέπει να αναγνωρίσουμε, ιδιαίτερα όταν εξετάζουμε τις μελλοντικέ εμπορικές συμφωνίες, είναι το γεγονός ότι για πολλές φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες μια τέτοια συμφωνία είναι Ε, για μας η δεύτερη καλύτερη λύση, όμως αυτοί προτιμούν τις διμερείς συμφωνίες, γιατί έτσι μπορούν να διαπραγματευτούν και μπορούν να μιλήσουν για θέματα τα οποία είναι πιο λεπτά και ευαίσθητα για αυτούς. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε νομίζω. Έπειτα με ανησυχεί κάπως η παράγραφος 22 που λέει ζητά από την, από την Κομισιόν να επιβάλλει την πρόσβαση στην αγορά, νομίζω πως δίνει αυτό λάθο εντύπωση. Εντάξει, κάποιες φορές πρέπει να είμαστε σκληροί στι εμπορικέ διαπραγματεύσει, αλλά πρέπει να προσέξουμε το, την γλώσσα που χρησιμοποιούμε, γιατί έτσι ενθαρρύνονται αυτοί που είναι κατά των συμφωνιών αυτών. Δηλαδή μπορεί να τονίσουν τέτοιες ε, ε, παραγράφους. Έπειτα, μιλάτε για διάλογο ανάμεσα στους εμπορικούς εταίρους. Εγώ θα ήθελα να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό που μπορούμε να πετύχουμε από κοινού με άλλους εταίρους όταν πρόκειται για τον ΠΟΕ. Για παράδειγμα, θα ήθελα η Ένωση και η ΕΠΑ να δείξουν μεγαλύτερη πρωτοβουλία για θέματα όπως η Γεωργία, για παράδειγμα. Γιατί και οι δύο είμαστε ένοχοι για επιδοτήσεις της Γεωργίας. Ξέρω ότι είναι πολύ επίμαχο αυτό το θέμα και αντιφατικό, αλλά ή θα μπορούσαν ας πούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ ΕΕ να κάτσουν και να δούνε πώς θα προχωρήσει το θέμα και για ορισμένα από αυτά τα κομμάτια όπως η Γεωργία. Τώρα, μιλάτε για μέσα εμπορικής άμυνας και εδώ συζητάτε αυτό το θέμα είχαμε διάφορες εκθέσεις και στην περασμένη θητεία, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε νομίζω ότι αυτές οι συμφωνίες δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως προστατευτικά μέσα για να καλύψουν μη, ανταγωνιστικές, ε, ε, μη, ανταγωνιστικούς ε, κλάδους. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτόν τον περιορισμό. Και επίσης, τα μέσα εμπορικής άμυνας έχουν αντίκτυπο και στους ε, λιανοπολιτές αλλά και στους, πολιτές, στους αγοραστές που πολύ συχνά πρέπει να πληρώσουν το τίμημα. Καταπολέμηση της στόχιας. Έχετε δίκιο πως πρέπει να έχουμε μαζί μας τους πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών. Όμως, σε σχέση με το Ταμείο Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση, δεν θα ήθελα αυτό να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την αδυναμία κάποιων να προσαρμοστούν στην παγκοσμιοποίηση. Μήπως δηλαδή ενθαρρύνουμε έτσι τον κόσμο να μην βλέπει στο μέλλον, αλλά να προσβλέπει στην παρηγοριά ενός Ταμείου. Τελευταία μου παρατήρηση, θα πρέπει νομίζω να σκεφτούμε πιο δημιουργικά όσον αφορά την πνευματική διοκτησία. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει διαβάσει το βιβλίο του Chris Anderson που, λέει, που έχει τίτλο «Free», λέει ότι σε έναν κόσμο αυξημένων ε, δυνατοτήτων αποθήκευσης ε, αλλά και επεξεργασίας στο τέλος φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου πολλά ψηφιακά προϊόντα στον ψηφιακό κόσμο, τα περισσότερα προϊόντα καταλήγουν να είναι δωρεάν. Δηλαδή, οι εταιρείε οι ίδιε θα πρέπει να είναι πιο εφευρετικέ στον ψηφιακό κόσμο, γιατί βλέπουμε να, υπάρχει, να μην υπάρχει συνέχεια. Α πούμε, στην βιομηχανία τη μουσική, είπαμε, τώρα περάσανε στα MP3, ε, δεν φαντάζονταν τι εξελίξει. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ναι, μεν προστατεύουμε την πνευματική ιδιοκτησία, αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε πω οι επιχειρήσει θα είναι καινοτόμε και δεν θα κρύβονται πίσω από ένα παλιό φόρματ ή ένα παλιό επιχειρηματικό μοντέλο, να αναγνωρίσουν ότι πρέπει και αυτέ να αλλάξουν. Όχι μόνο στο ψηφιακό τομέα, αλλά και σε άλλου κλάδου. Αυτά. Και θα τα πω και με τον Ντάνιελ, ώστε να μην πλατιάσουμε πολύ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γκάσπερ για τα εντυπωσιακά και ενημερωτικά σχόλιά του. Και θέλω να πω ότι υποφελούμεθα στην Επιτροπή μας από τις ε, γνώσεις και του συναδέλφου δίπλα και υποφελούμεθα. Πρόκειται για ένα ευρύτατο θέμα. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να συγχαρώ και τον ε, κύριο ε, Σάκαρη που μας παρουσίασε ένα κείμενο τόσο συνοπτικό. Ίσως κάνω ένα σχόλιο που δεν είναι τόσο θετικό, αλλά πρόκειται για την πρώτη ε, ανταλλαγή απόψε. Δύο σχόλια θα κάνω. Στο τέλος της παραγράφου 38 σωστά υπογραμμίζεται πόσο σημαντικό είναι να προστατεύονται τα πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα ε, διατησίες. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και απασχολεί και κάποια εταιρεία που είναι στην εκλογική μου περιφέρεια που κάνει ε, αντιασφυξιογόνες μάσκες. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέγεται εδώ. Τα IPPR λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Άλλη μια παράγραφος στην οποία θα ήθελα, για την οποία θα ήθελα να είναι στον συνάδελφο. Είναι εκεί που γίνεται λόγος για τις ξένες αγορές δημοσίων συμβάσεων. Ξέρουμε ότι εδώ υπάρχει μια προσπάθεια όλα να γίνονται εν κρυπτό και παραβίστο. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δώσουμε το κατάλληλο να προσδώσουμε κατάλληλη σημασία που πρέπει να έχει ε, το άνοιγμα αυτό που αναφέρεται στις ξένες αγορές των δημοσίων συμβάσεων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον Ντάνιελ για την έκθεσή του σύντομο, εξαιρετικό και εύστοχο. Το κύριο θέμα εδώ είναι όταν τονίζεται, όπως στη σελίδα 5 εδώ, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ που το 2048 ε, του η ΑΕΠ τώρα βλέπουμε ε, να σύμφωνα με τις προβλέψεις το 2020 να έχουν πέσει ποσοστά αντίστοιχα 35 και 27. Αυτό είναι σημαντικό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες ζεμεύσεις και λιγότερη γραφειοκρατία σε όλες τις χώρες. Στη σελίδα 7 λέγεται ότι θα πρέπει να υπάρξουν και άλλου είδους ε, πολιτικές και λέγει ότι η εμπορική πολιτική δεν είναι αυτός ο σκοπός. Επίσης λέγεται εδώ, υπενθυμίζονται εδώ ποιοι είναι οι άλλοι τομεί πολιτική που πρέπει να ληφθούν υπόψη, τα δικαιώματα, εταιρική κοινωνική ευθύνη, περιβαλλοντική, πολιτική, αλλά και πάλι πιστεύω ότι στον εμπορικό τομέα βλέπουμε να υπάρχουν ακόμη περισσότερα προβλήματα σήμερα με την απώλεια θέσεων εργασίας και με τη στασιμότητα που επικρατεί. Σωστά λοιπόν λέγεται ότι λέγεται. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι εξαιρετική η έκθεση αυτή ως βάση συζήτησης για το θέμα αυτό το τόσο σημαντικό. που αφορά την εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στα πλαίσια στρατηγικής της Ευρώπης του 2020. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες, κάποια στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Θα μπορούσα ως παράδειγμα να αναφέρω την τις ε, απόψεις μας για τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Θεωρούμε στο Κοινοβούλιο ότι πρόκειται για την δεύτερη καλύτερη δυνατή αλλαγή λύση. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε κάποιες επικρίσεις, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι ακόμη και αν ακολουθήσουμε και μια άλλη προσέγγιση, δεν μπορούμε να απαλλαγούμε αυτές, διότι υπάρχουν θέματα τα οποία μόνον εκεί μπορούν να υπάρξουν συμφωνίες. Γι' αυτό γίνονται διαπραγματεύσεις τέτοιου είδους Ίσως θα έπρεπε λοιπόν να κάνουμε λιγότερες επικρίσεις, εάν βεβαίως γίνονται για να υλοποιούν τους στόχους για τους οποίους προβλέπονται. Τώρα, για τη ε, σχέση μεταξύ της συμφωνίας της εμπορικός και του κοινωνικού πτυχής. Ορισμένοι πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για τις εμπορικές συμφωνίες. Εγώ αντιθέτως πιστεύω ότι αν το, η κοινωνική πτυχή αφαιθεί κατά μέρος, δεν θα πηγαίνουμε σωστά. Πιστεύω αντιθέτως ότι θα πρέπει να αποτελούν μέρος όλων αυτών των εμπορικών συμφωνιών. και οι τέτοιου είδους συμφωνίες πιστεύω ότι θα πρέπει να ανοίγουν το δρόμο για βελτίωση των ε, κοινωνικών ε, συνθήκων. Αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε σε εμπορικού μας εταίρους. Βελτίωση των συνθήκων, των ανθρώπινων δικαιώματα και των κοινωνικών συνθήκων. Τρίτη παρατήρηση που θέλω να κάνω, η αμοιβαιότητα. Συμφωνώ με τις παραγράφους 24 και 25. Διερωτώ με όμως αν δεν θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδεξοι. Πρόσφατα δημοσιεύθηκε μία επιστολή που απέστειλαν και υπέγραψαν πολλά μέρη κυβερνήσεων της Γαλλίας, της Πορτογαλίας, της Γερμανίας για να ε, μιλήσουν περισσότερο για την αμοιβαιότητα και την αρχή της η οποία θα πρέπει να ισχύει και αυτά στις διάφορες εμπορικές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ των διαφόρων χωρών, ακόμη και των πιο διγμένων. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή την ιδέα της ε, ε, διεύρυνση τη αρχής τη εφαρμογή τη αμοιβαιότητα θα πρέπει να τονίσουμε περισσότερο. Τελικά πιστεύω ότι ότι πολλές φορές το θέμα των διαφορών και των συναλλαγματικών διαφορών μπορούν ίσως να χρησιμοποιηθούν και αυτό είναι κάτι το οποίο αποσιωπούμε πολλές φορές σαν μια κρυφή επιδάτηση των εξαγωγών από κάποιους. Αλλά αυτό πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε στις ε, εμπορικές συναλλαγές, συμφωνίες. Διότι μπορεί να οδηγήσει λανθασμένους κανόνες του παιχνιδιού. Εν πάση περιπτώσει, ακούστηκαν και οι απόψει των συναδέλφων. Πιστεύω ότι λαμβάνοντα αυτά υπόψη, ο συζητή θα κάνει στο τέλο μια εξαιρετική έκθεση που θα αντικατοπτρίζει τι απόψει όλη τη Επιτροπή. Θέλει κανεί άλλο να κάνει κανένα σχόλιο. Ξέχασα την Επιτροπή. Εάν θέλει να προσθέσει κάτι κάποιο εκ μέρου τη Επιτροπή. Ο Μιγγέλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου που συνέβαλαν στην σύνταξη της έκθεσης αυτής. Οι παρατηρήσεις είναι πολύ καλές. Θα μπορούσα να αφαιρθώ στα πρώτα σχόλια που έκανε ο εισηγητής όσον αφορά το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προσφέρει μακροπρόθεσμες προοπτικές. Κοιτάξτε, στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως το είπατε κι εσείς, αναφερόμαστε σε μια μακροπρόθεσμη εμπορική πολιτική οι σπόροι που σπέρνουμε σήμερα ουσιαστικά θα αποδώσουν καρπού σε 10, 20, 30 χρόνια. Επομένως, η πολιτική την οποία προτείνουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφέρει αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Η πρόταση φαντάζομαι βέβαια του εισηγητή είναι να έχουμε κάποιες οικονομικές μακροπρόθεσμε προοπτικές. Ως προ αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε διμερή αλλά και πολυμερή συμφωνία και διαπραγμάτευση κάνει μελέτες αντικτύπου μακροπρόθεσμες και χρησιμοποιεί μακροπρόθεσμες προβλέψεις εκτιμώντας τον αντίκτυπο που θα έχουν οι διαπραγματεύσεις αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους Ευρωπαίους δηλαδή παραγωγούς καταναλωτές και πολίτες αλλά και στην χώρα εταίρο. Καλύπτουμε κατά αυτόν τον τρόπο όλους τους τομείς, τη βιομηχανία, τη γεωργία, τις κοινωνικές πτυχές. Δεν κάνουμε βέβαια κάτι τέτοιο για τις χώρες με τις οποίες δεν διαπραγματευόμαστε. Μια επίσημη συμφωνία, για παράδειγμα, η Ηνωμένε Πολιτείε, η Ιαπωνία, Κίνα. Αυτή είναι πολύ σημαντική μας εμπορική εταίροι, αλλά Καταλαβαίνετε ότι οι προβλέψεις αυτές είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και δαπανηρές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να κάνει οικονομικές αναλύσεις για τους σημαντικούς αυτούς εμπορικούς εταίρους. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τους πόρους τους οποίους έχουμε αυτή τη στιγμή για να κάνουμε αναλύσεις των μικρότερων τρίτων χωρών με τις οποίες συνάπτουμε συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κάσπαρη, έχετε το λόγο για να κάνετε κάποιες τελικές παρατηρήσεις και να καταλήξετε σε συμπεράσματα για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που έκαναν παρατηρήσεις. Χαίρομαι ότι τις επόμενες εβδομάδες θα μιλήσουμε για τις... την βελτίωση του κειμένου. Ούτως ή άλλως εγώ, όπως μου υποδείξατε, θα ανατρέξω πραγματικές πληροφορίες για να εμπλουτίσω το κείμενό μου. Άκουσα την Κομισιό, αλλά λυπούμε που άκουσα επίσης ότι Η Κομισιό ανέφερε ότι θα πρέπει, δεν είδε ότι θα πρέπει να έχουμε ε, υπομονή και να οργανωθούμε, διότι αυτά τα οποία θα κάνουμε τίποτε θα αποφέρουν κέρδη για τα 20 επόμενα 30 χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν τα διάφορα διαφορετικά σενάρια να τα λάβουμε υπόψη, να τα φανταστούμε. Πρέπει να ξέρουμε τι πρέπει να περιμένουμε και πώς φανταζόμαστε τι θα είναι ο κόσμος μετά από 15-20 χρόνια. Αναφερόμαστε στις συμπορικές συναλλαγές με την Ινδία αλλά θα πρέπει να δούμε και εκτός από τα δικά μας τα συμφέροντα σήμερα ποια είναι και τα συμφέροντα των ε, εμπορικών μας εταίρων και να σκεφτούμε και πάλι επαναλαμβάνω πώς θα είναι ο κόσμος σε 15-20 χρόνια διότι η εμπορική μας πολιτική θα πρέπει να μπορέσει να προσαρμοστεί στις ανάγκες του μέλλοντος. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας την πολυτέλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είμαστε σε μία θέση παρατηρητού, να βλέπουμε τι θα συμβεί σε 15-20 χρόνια. Θα πρέπει να είμαστε πρωταγωνιστές των αλλαγών. Σας ευχαριστώ. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών, λαμβάνοντας υπόψη αυτό το οποίο είπε προηγουμένως ο εισηγητής, 24 Μαρτίου. Εκπνέει προθεσμία στι 24 το μεσημέρι, 12 το μεσημέρι. Αντί 18 λοιπόν, αλλαγή για τις 24. Παρατείνεται λοιπόν η προθεσμία κατάσταση τροπολογιών κατά μία εβδομάδα. Το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη. 32. Τροποποίηση του κανονισμού περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μετασφοράς, της μεσητής και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης. Εγώ είμαι ο εισηγητής και επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για το θέμα αυτό. Το σύστημα που αφορά την εξαγωγή των ε, ε, προϊόντων και ειδών διπλής χρήσης μιλά περί κανονισ... αφορά κάποιες αλλαχές. Εδώ ε, αναφερόμεθα στην τροποποίηση των ε, παραρτημάτων που αφορούν κυρίως κάποια είδη διπλής χρήσης στην οποία περιλαμβάνονται προϊόντα και αγαθά και τεχνολογίες διπλής χρήσης για συμβατικά όπλα κτλ. Στο άρθρο 15 του κανονισμού προβλέπεται ότι ο κατάλογος αυτών των ειδών διπλής χρήσης θα πρέπει να ενημερώνεται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και τροποποιήσεις αυτών που έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη ως συμβαλόμενα μέρη των οικείων διεθνών καθεστώτων μη διάθεση και διευθετήσεων ελέγχου των εξαγωγών με την κύρωση των οικείων διεθνών συνθήκων. Η τελευταία επικαιροποίηση του παραρτήματος πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία τη έκδοση του κανονισμού στις 5 Μαΐου 2009. Από τότε όλα τα διεθνή συστήματα ελέγχου των εξαγωγών έλαβαν την απόφαση να τροποποιήσουν και να επικαιροποιήσουν τους κατάλογους και να κάνουν απαραίτητες απαραίτητε του παραρτήματος 1. Έχει φτάσει σήμερα στο Κοινοβούλιο η πρόταση της Επιτροπής για τις τροποποιήσεις. Εμείς έχουμε πολύ μικρό περιθώριο ελιγμών. Έχουν υπάρξει συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών και το παράρτημα θα τροποποιηθεί. Θα πρέπει να γίνουν οι διάφορες αλλαγές. Ε, το έγγραφο τροποποιείται, υποβάλλεται στα κρατημέλη, τα οποία πρέπει να κάνουν σχόλια. Το θέμα τα συζητείτε και πάλι όταν επανέρχεται στο Συμβούλιο, όταν συμφωνήσει με τροποποίηση του παραρτήματος το Συμβούλιο, το μεταφράζει το έγγραφο στις επίσημες γλώσσες, το σχέδιο στέλνεται μεταφρασμένο έτσι ως έχει στην Επιτροπή. Οι προτάσεις αυτές αποτελούν νομοθετική πρόταση που αποβάλλει η Επιτροπή ελέγχει όλες τις διαδικασίες και στο τελικό σχέδιο εγκρίνεται η πρόταση και την αποστέλει και πάλι στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Βλέπετε λοιπόν ότι η διαδικασία είναι πολύ πολύ πολύπλοκη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει την δυνατότητα να τροποποιήσει την όλη διαδικασία ως θεσμικό όργανο. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να αναφερθούμε. Αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε, μάλλον θα ακολουθήσει ένα τριμέρη διάλογος με το Συμβούλιο για την πρόταση κανονισμού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για να τροποποιηθεί ο κανονισμός 34 του 2000 που θα δημιουργεί ένα κοινοτικό καθεστώς για το καθεστώς εξαγωγής ειδών διπλής χρήσης εδώ καταφέραμε να πετύχουμε σημαντικές τροποποιήσεις στο άρθρο 1 του κανονισμού αυτού. Πιστεύω ότι αυτές τις τροποποιήσεις θα πρέπει να υπερασπιστούμε. Αν χρειαστεί να εγκρίνουμε πολύ γρήγορα το παράρτημα υπαριθμών 1, θα μπορούμε τουλάχιστον να χρησιμοποιήσουμε ως διαπραγματευτικό χαρτί τις τροπολογίες οι οποίες έχουμε υποβάλει για τις τρεις προηγούμενες εκθέσεις. Γι' αυτό λοιπόν σας προτείνω στο παράρτημα υπαριθμών 1 του κανονισμού αυτού να συμπεριληφθούν και οι τροπολογίες αυτές που είχαμε υποβάλει για τα προηγούμενα νομοθετήματα. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποια είναι η αποψή σας για το ζήτημα αυτό. Θα ήθελα να μου πείτε και αν συμφωνείτε λοιπόν με την πρόταση αυτή, αν αξίζει να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Και θέλω βέβαια και τη δική σας έγκριση προτού υποβάλλω το σχέδιο έκθεσης. Δεν έχουμε πάρα πολλά μέλη αυτή τη στιγμή στην αίθουσα. Σας ακούσουμε λοιπόν τον Πάολο Γκαρτζότη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, τον κύριο Ριτσκόφσκι. Συγγνώμη για τον τρόπο που πρόφερα το όνομά σας. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετική η παρουσίασή σας, επομένως δεν θα επαναλάβω αυτή τη στιγμή τα όσα άλλωστε λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έγγραφο. Θα αναφερθώ σε ένα-δύο σημεία τα οποία αξίζει να τονίσουμε. Πρώτον, ο λόγος για τον οποίο γίνονται κάποιες τροποποίησεις όσον αφορά το παράρτημα 1, τον κατάλογο ελέγχου εξαγωγών. Τρεις βασικούς λόγους έχουμε τεχνολογική πρόοδος, δεύτερον η διαθεσιμότητα κάποιων ειδών, καθώς επίσης και τρίτον κάποιες νέες ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια, ανησυχίες που έχουν ορισμένα κράτη και τα οποία, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Έτσι λοιπόν στον κατάλογο που έχουμε στο παράρτημα επικαιροποιούνται εδώ πέρα τα στοιχεία προκειμένου να καταφέρουμε να ευθυγραμμιστούμε περισσότερο με τις παγκόσμιες εξελίξεις όσον αφορά τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα νέα αυτά είδη τα οποία παρουσιάζονται. Η πρόταση που έχετε μπροστά σας όσον αφορά την τροποποίηση του καταλόγου αυτού ελέγχου στο παράρτημα 1 διαφέρει από τις υπόλοιπες προτάσεις που έχετε πάλι μπροστά σας όσον αφορά τις γενικότερες αδειοδοτήσεις εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι υπάρχει ένας μικρός κινδύνος επικάλυψης εδώ πέρα. Οι άλλες ε, προτάσεις που έχουν να κάνουν με το γενικότερο καθεστών εξαγωγών έχουν να κάνουν μόνο με τις κατηγορίες των ειδών που επικαιροποιούνται στο παράρτημα 1. Ακόμα και γίνονται λοιπόν κάποιες αλλαγές στο παράρτημα υπαριθμών 1 οι ε, γενικές άδειες τις οποίες ε, εξετάζουμε θα λάβουν αυτόματα υπόψη τους και τις αλλαγές αυτές και κατά αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί η εξαγωγή των ειδών αυτών προς τρίτες χώρες. Μια τελευταία τώρα παρατήρηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται μια νέα πρόταση που θα υποβληθεί στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπάρχει μια επιταχυμένη διαδικασία τροποποιήσεων των τεχνικών αυτών παραρτημάτων των μελλοντικών αλλαγών που θα γίνουν. Βέβαια, η πρόταση παραμένει ίδια εδώ. Ευχαριστώ. Particularly... Σας ευχαριστώ για τι παρατηρήσει σα. Όντω έπρεπε να γίνουν οι αλλαγές αυτές, να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος και να γίνουν αλλαγές. Ο κύριο Κάσπαρη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως και εισηγητής για την ομάδα μου, Βασικά συμφωνώ με τα όσα είπατε. Νομίζω ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει επικάλυψη Αν έχω ενημερωθεί καλά, δεν θα υπάρξει επικάλυψη και από τα όσα άκουσα από την ε, Κομισιόν πρόκειται μόνο για τα παρτήματα εδώ. Αλλά θα πρέπει να βαγιαστούμε νομίζω, γιατί αυτός ο κατάλογος, ε, ενημερωμένος κατάλογος θα έπρεπε ήδη να έχει εισαχθεί και θα πρέπει αυτό να γίνει όσο γίνεται πιο σύντομα να γίνει αυτό σύντομα χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο την έκθεση ε, αιστρία. Μάλιστα. Λάβουμε υπόψη και τα όσα είπε η Κομισιόν και θα προχωρήσω στην προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε τώρα το εξέταση μερικής διάταξης. Δεν έχουμε τίποτα στα διάφορα. Η επόμενη μας συνεδρίαση θα γίνει στις 12 και 13 Απριλίου. Εδώ στις Ρυξέλλες. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και για τη συνεργασία σας.